Well, good morning, everybody. I think um, uh, we can make a start on uh, our agenda for today because uh, we have big votes to come at 10 o'clock. Έχουμε ψηφοφορίες που ξεκινάνε στις 10. Ας περάσουμε στο πρώτο σημείο που είναι η δέσμη μέτρων ευθυγράμμισης για μια σειρά από σημαντικά μέσα για τα προϊόντα. Η κυρία Ρόιτοβα ε, διευθύνει την όλη διαδικασία και θέλουμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Θα το ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Διότι έχουμε άλλες σημαντικές ψηφοφορίες σήμερα το πρωί. Έχουμε την κυρία Σαλεμός εδώ από τους σοσιαλιστές και τον κύριο Μάντας. Η κυρία Ρούντ δεν είναι ακόμα εδώ. Ο κύριος Φόξ δεν είναι εδώ. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν μέσα στην πρώτη μισή ώρα. Διότι έχουμε και μία παρουσίαση ε, από τον κύριο Αέρας ε, στις 9.30. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Χαίρομαι που καλωσορίζω την κυρία Μπρίγκμαν και την ομάδα της από τη Γενική Διεύθυνση Enterprise ε, που είναι θεματοφύλακες αυτής της πρότασης που μας την έστειλαν για εξέταση. Επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει το μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας μετά από το έργο μας για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων η αγορά αναμένει τη νέα σας πρότασμα που θα αποτελέσει κομμάτι του προγράμματός μας για του χρόνου. Όλοι οι συναδέλφοι έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρώ ότι θα είναι μια από, τους, από τις πρώτες προτεραιότητες μας ως φάκελος. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα μετά από όλη τη δουλειά που κάναμε για τις υπηρεσίες να αρχίσουμε να μελετάμε και τα ζητήματα για τα εμπορεύματα. Το 2013 θα είναι το έτος για τα εμπορεύματα, για την ασφάλεια των αγαθών. ορίζουμε επίσης και το κρατηριό μας μέσω διαδικτύου, πολλοί άνθρωποι ε, από οργανισμούς τυποποίησης ε, και άλλες αγορές παρακολουθούν από απόσταση αυτή τη συνεδρίαση για να μας πείτε τις απόψεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστοτοπού μας και επίσης ε, μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό μας δελτίο online ε, που σας αναφέρει όλα τα θέματα τα οποία μελετάμε και σας παρέχει συνδέσεις για τα έγγραφα. Μπορείτε να βρείτε έτσι όλα τα έγγραφα για οτιδήποτε συζητάμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν έχουμε τίποτα ή κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Καλό λοιπόν την Ζωζάνα Ροϊτόβα να μας παρουσιάσει και να απαντήσει στις ε, ε, τροπολογίες που υποβλήθηκαν για την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους και συζήτητες και τους βοηθούς καθώς και τη γραμματεία για τη συνεργασία τους. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που επικοινωνούσε μαζί μας, συνεργάστηκε μαζί μας τόσο άμεσα. Αυτό το πακέτο ασχολείται με το marketing αγαθών, με την εμπορευματοποίηση αγαθών και όλες αυτές οι προτάσεις είναι ουσιαστικά σημαντικές. Όλες αφορούν την ευθυγράμμιση με τη δέσμη μέτρων για τα εμπορεύματα του 2008. Ε, υπάρχουν κάποιες νομοθετικές και κάποιες τεχνικές, ε, κάποια τεχνικά ζητήματα υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις για τη διαδικασία επιτροπολογίας. Δεν λάβαμε τη θέση για τα παρατεχνικά και, ε, μέσα. Καλό λοιπόν την Κυπριακή Προεδρία να ολοκληρώσει αυτό που πρέπει να γίνει. Συνολικά έχουν υποβληθεί 500 τροπολογίες περίπου συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπήρχαν στις εκθέσεις μου. Θα εστιαστώ σε τέσσερις τομείς. Το ζήτημα της νομικής βεβαιότητας, επίσης της προστασίας των καταναλωτών και μετά το να βεβαιωθούμε ότι θα απαλείψουμε το διοικητικό φόρτο και την γραφειοκρατία για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Επίσης, να διαβεβαιωθούμε, να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρχει θέμα του ανταγωνισμό. Έχω προτείνει έξι οριζόντιες τροπολογίε, συμβαστικέ και μία τομεακή. Μία για τα όρια τάση. Έχουμε συγχωνεύσει κείμενα. Όσον αφορά το ερώτημα του κατά πόσο η απεικόνηση, η εικόνα ενός ε, προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνεται στο DLC. Η οριζόντια συμβαστική τροπολογία επίσης διασαφενίζει ορισμένα σημεία τα οποία σχετίζονται με τους διανομής και τις αποθήκες εμπορευμάτων μετά από την υιοθέτηση των νέων κανόνων και την υλοποίησή τους και την εφαρμογή τους. Αυτό θα σημαίνει απαγόραυση οποιασδήποτε ε, δρομικής εφαρμογής. Αυτό ισχύει επίσης για κάποια δεδομένα αναγνώρισης στις συσκευασίες και στα έγγραφα. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι εύκολο να κατανοηθούν από τους καταναλωτές και από τις εποπτικές αρχές. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ταχυδρομική διεύθυνση ενώ η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε πρώτα για τα απλά δοχεία πίεσης με την υιοθέτηση την απόρριψη των οριζόντιων ε, συμβιβαστικών τροπολογιών ε, θα εφαρμόσουμε το ίδιο και στις υπόλοιπες έξι Αναφερόμενοι τώρα σε συγκεκριμένες τροπολογίες, η συνάδελφος Φερμπόντ έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο. Δεν εγκρίνω την πρότασή της να προβλέψουμε υποχρεωτικό DLC για κάθε προϊόν, διότι αυτό θα κόστιζε υπερβολικά πολύ. Όσον αφορά το υποχρεωτικό σύστημα διαπίστευσης, εδώ προτιμώ να προτιμώ να υποστηρίξω την Κομισιόν και το σχέδιο της αναθεώρησης αυτής της δυνατότητας και τη μελέτη αντικτύπου. Θα Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή έχει εκφράσει την άποψή της γι' αυτό όσον αφορά την άποψη του Συμβουλίου είναι και αυτή αρνητική. Υποστηρίζω τις τροπολογίες για να επανέλθω στον ορισμό, στον τυπικό ορισμό των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών επειδή μας παρέχει ε, περισσότερη βεβαιότητα όσον αφορά την Ερμηνεία. Επιπλέον υποστηρίζω επίσης ε, τη χορήγηση εξαίρεση συγκεκριμένα για εμπορεύματα που προορίζονται για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς μόνο. Όσον αφορά τις πληροφορίες ασφαλείας, αυτές θα πρέπει να είναι εύκολες στην κατανόηση και σαφείς. Κάποιοι έχουν λάβει κείμενα ε, από παλιά έγγραφα και αυτές οι διατάξεις ουσιαστικά δεν περιλαμβάνουν κάποια μεγάλη αλλαγή ή κάποιες μεγάλες επενδύσεις. Όσον αφορά την πρόταση για κάποιες ευάλωτες ομάδες καταναλωτών, Εδώ βασιστήκαμε δειγματοληπτικά σε κάποιες διατάξεις που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Έτσι παρέχεται ένα ισορροπημένο πλαίσιο και όπως ακριβώς ο όρος για την εύλογη χρήση αυτών των εμπορευμάτων στο πλαίσιο των απαιτήσεων ασφαλείας όπως προβλέπονται στον 735 καθώς 2008. Καθώ θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε επίση και τι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι επιστημονικέ και τεχνικέ διαβουλευσει. αναμένω να συνεργαστώ με την Κυπριακή Προεδρία και θα ήθελα να μας εξηγήσουν Ποιο είναι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα για όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματίες μας θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο όλες αυτές τις αλλαγές. Εάν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνέψει αυτή τη συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, είμαι διατεθειμένη εφόσον γίνει αυτό στο πρώτο τρίμηνο του φθινοπόρου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τον Ιούλιο ή στις αρχές Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο θα πρέπει να παρουσιάσει μια θέση. Ευχαριστώ. Good. Thank you. πολύ ωραία. Σας κάτι ευχαριστώ. Είναι κανείς εδώ από την Κυπριακή Προεδρία. Α, ναι, ναι, ναι. Η Μαρία. Μήπως αργότερα να μιλήσει. Ε, συγγνώμη, δεν σε είχα δει πριν γιατί συνήθως το Συμβούλιο κάθεται μπροστά από την Κομισιόν, αλλά έχει αλλάξει η διευθέτηση φαίνεται. Είπα ξανά ότι σας κατευχαριστώ για όλες σας τις προσπάθειες σε αυτό το τόσο πολύπλοκο θέμα. Τώρα θα ακούσουμε τους σκιώδεις και τις σκιώδεις. Η κυρία Σάλντε Μόζερ πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Ρόιτοβα. Οι διαπραγματεύσεις μας ήταν πολύ θετικές και τα πράγματα δύσκολα. Υπήρξε ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας για ώστε να επιτευχθεί μια σωστή λύση αυτό υπήρξε θεμελιώδη σημασία. Ήταν επίση σημαντικό αυτή η διαδικασία να είναι μια διαδικασία ευθυγράμμιση. Λαμβάνουμε υπόψη και την απόφαση του 2008 τη δεσμή μέτρων για τα εμπορεύματα. Ήταν μια εξαιρετικά ορθή απόφαση. Γι' αυτό το λόγο οι οδηγίε προσαρμόστηκαν στι αποφάσει εκείνης τη εποχή. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να ξανανοίξουμε αυτό το πλαίσιο και να προσθέσουμε νέε πτυχέ υπερβολικά πολλέ νέε πτυχές. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει μια εξαιρετική ισορροπία σε αυτό το επίπεδο. Αν τώρα εγκριθεί σήμερα, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε μια πιο ασφαλή εσωτερική αγορά, αλλά και πιο αποτελεσματική, που θα λειτουργεί καλύτερα χάρη σε όλες τις οδηγίες που τίθενται σε ίσχυ. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, η ομάδα των σοσιαλιστών υποστηρίζει την πρόταση που σχετίζεται με το υποχρεωτικό σύστημα διαπίστευσης. Ωστόσο, δεν είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να το προσθέσουμε τώρα στην οδηγία. Πρέπει να περιμένουμε τη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν, αλλά πιστεύουμε πιο μακροπρόθεσμα σκόπιμο θα ήταν να προσθεθεί. Μετά, όσον αφορά το γεγονός ότι όλη η παραγωγή Όλοι οι κατασκευαστές ε, πρέπει να επισυνάπτουν μια δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντο με τους κανόνες. Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις με αυτό το διοικητικό φόρτι, με αυτή την υποχρέωση δήλωσης. Ε, δεν είναι αποφασιστικός παράγοντας αυτή η δήλωση οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να παίρνουν αυτή την δήλωση εφόσον το ζητήσουν. Δεν χρειάζεται σόνι και καλά να επισυνάπτεται στα εμπορεύματα. Κατά τα άλλα, όπως έλεγα, είμαστε πεπισμένοι ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η εσωτερική αγορά, θα λειτουργεί καλύτερα και θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας και περιμένουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστούμε. Uh, thank you very much, Mr. Και εσάς σας ευχαριστώ κύριε Σαλντεμόζερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω θα καταθέσει προφορική τροπολογία η κυρία Σαλντεμόζερ. Δεν ήμουν σίγουρη γι' αυτό το ρωτάω. Κατά τα υπόλοιπα φαντάζομαι ότι Αυτά που είπε η Κομισιόν για την ασφάλεια των προϊόντων ισχύουν. Συμφωνώ εδώ με την κυρία Ροϊτόβα ότι δεν πρέπει να, να γράφει αυτά στην οδηγία. Απλώς να γίνει η μεταφορά της δέσμης για τα εμπορεύματα χωρίς τίποτε παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάντως γενικά για τη συνεργασία μας και τους συμβιβασμούς που πετύχαμε. Θα τα υποστηρίξουμε όλα αυτά στην ψηφοφορία. Μήπως η κυρία Σαλτεμόζερ να επανέλθει αργότερα. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φόξ και μετά θα συζητήσουμε αυτά που είπε η κυρία Ρούλε, κύριε Φόξ. Ευχαριστώ την κυρία Ρόιτοβα και τις υπηρεσίες του συνεργάτες της. Η ομάδα μου μπορεί να υποστηρίξει τους περισσότερους συμβιβασμούς και τις τροπολογίες των συναδέλφων που διορθώνουν ορισμένες ελλείψεις της αρχικής πρότασης και που ελαφρύνουν κάποια βάρη που πρόσθεταν στις επιχειρήσεις. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω την αλλαγή της τροπολογίας που έχει καθοριστεί από την οδηγία και προτείνω να αντικατασταθεί η λέξη όργανο ή εργαλείο με τη λέξη apparatus. Ελπίζω αυτό να το δέχεται η συγγήτρια και οι συνάδελφοι. Ελπίζω να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση της κυρίας Ροϊτόβας. Α, ευχαριστώ για την τόσο λεπτομερή σας εργασία. Πρώτα το ερώτημα της κυρίας Μόζερ και μετά θα επανέλθουμε στην κυρία Ρόιτοβα. Τα λέω αγγλικά για να είναι σαφέστερα τα πράγματα. Λοιπόν, οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν την προσέγγιση της κυρίας Ρόιτοβας δηλαδή. Συμφωνούμε με τις ιδέες think... της κυρίας Βανούς. Με βάση την αξιολόγηση της Κομισιόν. Γι' αυτό δεν θα καταθέσουμε ούτε προφορικές τροπολογίες ούτε τίποτε άλλο. Όσο για την υποχρεωτική επισύναψη αυτή αυτών που προτείνει η κυρία Ρόιτοβα θα συνεννοηθούμε ξανά και θα δούμε. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοούσα γιατί τα είπα αγγλικά. Ε. Ναι, ναι, μα πράγματι πολύ λογική αυτή η πρόταση. Γιατί θα μας ξανάρθει το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων και του χρόνου. Μήπως κανείς άλλος ή καμία άλλη θέλει να σχολιάσει. Όχι, κυρία Ρόιτοβα. Μήπως να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και το Συμβούλιο όμως. Κυρία Μπρίνκμαν να σχολιάσει τις τροπολογίες και μετά και η Δανική Προεδρία λέει ο Πρόεδρος. Α, όχι η Κυπριακή, η Κυπριακή. Είναι πρώτη φορά που έρχεται, γι' αυτό ότι καλωσορίζουμε θερμά. Ναι, ναι, η Κυπριακή, η Κυπριακή Προεδρία. Λοιπόν, πρώτα όμως η κυρία Μπρίνκμαν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ρόιτοβα για τη σκληρότατη εργασία που προφανώς χρειάστηκε να κάνει για αυτή την σημαντική πρωτοβουλία και ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Επομένως, οι περισσότερες τροπολογίες που θα ψηφιστούν το απόγευμα, λέει ο Μιλήτρια, είναι μια πραγματική απτή βελτίωση του αρχικού κειμένου της οδηγίας και οι συμβιβαστικές δείχνουν τι σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για να καταλήξουμε εκεί. Βεβαίως λογικό θα ήταν να αναμείνουμε λογικό ήταν που συζητήθηκαν τόσο πολύ ορισμένα θέματα αν και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στην οδηγία γιατί ξεπερνούν το εύρος της, το θέμα της Θα ήθελα όμως να πω ότι η Κομισιόν θα κάνει ευρεία διαβούλευση για την εσωτερική αγορά βιομηχανικών προϊόντων του χρόνου και εκεί θα, υπά, θα δοθεί ένα βήμα για τη συζήτηση των βασικών στοιχείων της προσέγγισης μας και ορισμένων από τα πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν εισαγωγές από τρίτες χώρες και το κατά πόσον θα έπρεπε αυτή η πιστοποίησή τους να είναι υποχρεωτική ή όχι. Είναι βέβαια απογοητευτικό ότι τα εργαλεία μέτρησης προσωρινά ελπίζω έχουν διαγραφεί από τη δέσμη που θα ψηφιστεί το απόγευμα, αλλά πιστεύω ότι το αδιέξοδο αυτό θα μπορέσει να λυθεί για να μπορέσουν και οι δύο οδηγίες να εγκριθούν ίσως το Σεπτέμβριο. Κρίμα θα ήταν να έχουμε φτάσει μέχρι αυτού του σημείου και τελικά να διαλυθεί η συνδυασμένη πρόταση των τριών μέτρων αφού μπορεί να υπάρξει συνεννόηση πριν λήξει το έτος. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου θα καταλήξει σε αίσιο τέλος και θα ωφελήσει όλους τους οικονομικούς παράγοντες και τις αρχές των κρόνων μελών. Καταλήγω λοιπόν ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους σας που με, τόση, με τόσο πνεύμα πρωτοβουλίας και θέλησης κατέληξαν στους συμβιβασμούς που θα ψηφίσουμε σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Μπρίνκμαν μου. Η κυρία Τσιγκού από την Κυπριακή Προεδρία να μας πει δύο λόγια γιατί προεδρεύει τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου σχετικώς. Ξέρω ότι οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου εξετάζουν αυτό το δεύτερο ή τρίτο θέμα που ανέφερε η εκπρόσωπος της Κομισιόν και πέστε μας και εσείς δύο λόγια. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Πρόεδρέ μου. Ευχαριστώ και την κυρία Ρόιτοβα με τους συνεργάτες της. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν το έργο της γιατί είναι πολύ τεχνικό το θέμα. και πρέπει να τη συγχαρούμε. Η Κυπριακή Προεδρία έχει ήδη αρχίσει την επεξεργασία του θέματος και θα επιταχύνει ώστε να καταλήξει σε κάποια θέση που να σας την παρουσιάσει το Σεπτέμβριο. Όσο για τα δύο συγκεκριμένα άλλα θέματα που αναφέρατε, ελπίζω η διαφωνία μεταξύ ημών και της νομικής υπηρεσίας να μην συνεχιστεί και να μην αποτελέσει φραγμό στην πρόοδο των εργασιών μας. Ελπίζουμε δηλαδή να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να βρεθεί μια κομψή λύση για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα της επιτροπολογίας που λένε γιατί και η βιομηχανία αναμένει πρόοδο. Βιομηχανία. Μάλιστα, η διαμάχη μεταξύ νομικών υπηρεσιών είναι κάτι το τρομακτικό. Ίσως να μπορέσουμε τελικά να προσπάσουμε κάποια λύση και εσείς μηχανικός είστε κάτι θα καταφέρετε. Θα δούμε οι δικηγόροι τι θα κάνουν. Λοιπόν, η κυρία Ρόιτοβα. Ρόιτοβα. Θα ήθελα και εγώ να επιστήξω ότι όντως θα είμαι υπέρ των ε, προφορικών τροπολογιών που κατατέθηκαν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ε, συμφωνίας που αφορά την ε, ε, την διαπίστευση θα περιμένω να αποφασίσει η Επιτροπή ποια θα είναι το αποτέλεσμα στο οποίο θα κατελήσει. Τώρα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ έκανα κάτι το παρεμφερές όσον αφορά τα συστήματα υγείας και ξέρω περί των Τώρα, όσον αφορά την Κυπριακή Προεδρία, άκουσα με ευχαρίστηση ότι πρόκειται για ένα θέμα προτεραιότητα και θα ήθελα να πω ότι και εγώ και οι σκιώδεις συζητητέ συμφωνήσαμε ότι οι τροπολογίε, οι οποίες είναι οριζόντιε και για τις 7 ε, οδηγίες θα παραμείνουν και για τις δύο τις οποίες δεν θα ψηφίσουμε. Κατάλαβα ότι έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά περί τίνος πρόκειται η Κυπριακή Προεδρία και όντως θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους σαφείς κανόνες για όλους τους κατασκευαστές ό,τι και να κατασκευάζουν. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε, όπως είπατε όλοι, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε κυρίως τον βοηθό μου για την δουλειά που έκανε και ξέρω ότι πολλές φορές όταν ε, συνεργάζονται και γιατροί και δικηγόροι, ε, όλα πάνε καλά. Ε, χρειάζεστε και λίγους μηχανικούς εκεί και όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε ότι θα ψηφίσουμε τις 7 οδηγίες με και τις δύο εναπομένες το συντομότερο δυνατό. και βεβαίως για την ασφάλεια των προϊόντων και την επιτήρηση των αγορών θα συνεργαστούμε, ελπίζω, πολύ θετικά με την Κομισιόν για να περάσουμε και τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα είναι το κυρίου Αρίας, τον οποίο περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα έρθει όσο να κύριος Αρίας θα μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονόριο. Παρακολουθήσαμε διάφορες συναντήσεις, διότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ξέρουμε ότι παρακολούθησε και το... Και επειδή ήταν δημόσιες συνεδριάσεις, παρουσιάστηκε μεγάλο ενδιαφέρον και εκ μέρους των ε, καταναλωτών και επίσης πρέπει να πω ότι οι οργανώσεις καταναλωτών για αυτά τα θέματα επίσης μας παρουσίασαν ιδέες για θέματα ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στον τομέα αυτό. Και επίσης από το λιανικό εμπόριο είχαμε πολλές συνεισφορές. Engaging the retail sector more deeply in our own work on the single market.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 Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στον τομέα του λιανικού εμπορίου και επειδή αλλάζουν τα πράγματα, πολλοί με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν να καταλήξουμε εμείς στα πλαίσια της ενιαίας συντορικής αγοράς σε συμπεράσματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσπιζόμαστε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα και σίγουρα μας αναμένουν τα αποτελέσματα. τυπωσούνται με το λιανικό από τις συζητήσεις που έγιναν χθε, σε μια συζήτηση που είχα εγώ με το Eurocommerce, κατάλαβα ότι, σύμφωνα με αυτό που είπε η Επιτροπή, ελπίζουν ότι θα υπάρξει και μία πράσινη βίβλος για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως για την παράδοση πακέτων. Ξέρουμε ότι πολλά προβλήματα τα οποία έχουν οι καταναλωτές έχουν να κάνουν με την δυσπιστία που έχουν όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Διότι δεν ξέρουν αν τελικά ένα προϊόν το οποίο παρήγγειλαν θα φτάσει στα χέρια τους, αν θα τους αρέσει, πώς θα το επιστρέψουν, αν δεν ε, πάει κάτι καλά. Όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τις ε, συναλλαγές στο ηλεκτρονικό ελληνικό εμπόριο τους ενδιαφέρουν. και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, οι περιορισμοί που τίθενται, διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να λειτουργήσει η ενιαία εσωτερική αγορά. Επίσης, ξέρουμε ότι ε, στην Γερμανία υπάρχει το πρόβλημα του υψηλού κόστους παράδοσης κατοίκων αυτών των προϊόντων. Η ενιαία λοιπόν ψηφιακή αγορά έχει προβλήματα. Μίλησα εγώ για όλα αυτά τα προβλήματα πριν να έρθετε κυρία Ρίας. Έκανα το ζέσταμα, όπως λέμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού ήρθατε, εσείς έχετε το λόγο τώρα. Έλεγα, λοιπόν, ότι η δουλειά η οποία έγινε στο ομάδα εργασία μας βοήθησε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και μέχρι τις 10 που είναι ώρα ψηφοφορίας θα σας ε, δώσω τον λόγο να μας μιλήσετε, να γίνουν ερωτήσεις ε, θέλετε, χρειάζεστε οθόνη, θα παρουσιάσετε διαφάνειες, όχι, σας δίνω αμέσως το λόγο για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας και μετά υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη που θέλουν να συνεισφέρουν στη συζήτηση, θα του δώσουμε το λόγο. Έχετε το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου. Γιατί τον προηγούμενο μήνα έπαθα κάποιο ατύχημα και δεν μπορώ να τρέξω. Έτσι λοιπόν ήρθα με λίγη καθυστέρηση. Μαύρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα τη Ομάδα Εργασία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την ενιαία ψηφιακή αγορά. Αρχίσαμε πέρσι στι 11 ε, Ιανουαρίου σε αυτό το δεύτερο κύκλο. Είχαμε 7 συνεδριάσεις, μία κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήσαμε πολλά θέματα όπως και στις προηγούμενες του πρώτου κύκλου. Σε αυτές λοιπόν τις συνεδριάσεις λύσαμε να διατηρήσουμε τον ίδιο στόχο και το ίδιο πνεύμα όπως και πέρσι. Δηλαδή να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ανοιχτή βάση συζήτησης, μελέτησης και ε, ανάλυσης όπου εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και κάποιοι από τους περισσότερους εμπλεκόμενους σημαντικούς φορείς να παρουσιάσουν την κατάσταση για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή αγορά για να μπορέσουμε να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις και να κάνουμε προτάσεις για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Σε κάθε συνεδρίαση προσπαθήσαμε από μία ε, με ανοιχτό τρόπο να ασχοληθούμε με τα διάφορα θέματα και προσπαθήσαμε να ακούσουμε τις περισσότερες δυνατές οπτικές γωνίες ώστε να έχουμε μία ε, ευρεία προσέγγιση του θέματος. Πιστεύω τελικά ότι η ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση είναι κάτι το θετικό και μπορούμε μετά τη συζήτηση να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των θεσμικών οργάνων μας βοηθά στο να γνωρίσουμε και να παρακολουθήσουμε περισσότερο τα προβλήματα που γίνονται. Ως νομοθέτες, και την άποψή μου, νομίζω ότι θα πρέπει να ακούμε με προσοχή όλους τους ενδιαφερομένους και ε, να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις γνώσεις που γίνονται ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε τους καλύτερες δυνατές λίστα υπάρχοντα προβλήματα και για να ανταποκριθούμε περισσότερο και καλύτερα στις προκλήσεις αυτής της νέας τεχνολογικής εποχής μας. Με τον σαφή στόχο να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα μια ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Αφενός αναλύσαμε και συζητήσαμε τα θέματα της ε, πολιτικής ατζέντα των θεσμικών οργάνων δεδομένου ότι όλα αυτά έχουν ε, αντίκτυπο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Λάβαμε υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής και το, νομισματικό, ε, το, το νομοθετικό πακέτο για τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Επίσης ασχοληθήκαμε με θέματα τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι σημασίας, όπως ο ρόλος των ΜΜΕ και των λιανοπολιτών, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η εγγύηση προς τους καταναλωτές και να δούμε πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε το κατάλληλο πλωστάσιο στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην σωστή κατεύθυνση. Και θα, ε, δύο σημαντικά, θα αναφερθώ σε δύο σημαντικά θέματα. Στην ηλεκτρονική ε, ε, υπογραφή και στις ηλεκτρονικές συμβάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους τους συναδέλφους σας που συνεισέφεραν σημαντικά στην ε, συζήτηση και στην ε, εκπόνηση προτάσεων χρήσιμων, καθώς και για τη συμμετοχή τους συζητής. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξηγούσαν κατά την διάρκεια των συζητήσεων ποιες ήταν οι διαφορετικές προτάσεις που είχαν υποβάλει και απαντούσαν στις απαντήσεις που έκαναν όλοι οι συμμετέχοντες, εμπλουτίζοντας τον τρόπο αυτό όλες τις συζητήσεις. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εμπλεκόμενους φορείς που συνεισέφεραν και παρουσίασαν τις απόψεις για τα διάφορα θέματα, καθώς και για τους πραγματογνώμονες οι οποίοι μας παρουσίασαν διεξοδικά τις μελέτες τις οποίες είχαν κάνει και τις οποίες χρησιμοποίησαμε για τη διάρκεια των συζητήσεων στις διάφορες συνεταιρίες. Θέματα όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, η προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, το ΦΠΑ, οι δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ε, υπογραφή και ο ρόλος των ΜΜΕ αναλύθηκαν ευρύτατα και παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που σε μεγάλο βαθμό μας βοήθησαν να κάνουμε το σχέδιο απόφασης το οποίο παρουσίασα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Προσπάθησε εκεί να συγκεράσω τις διάφορες απόψεις που παρουσιάστηκαν στην ομάδα εργασία και τις προτάσεις που έγιναν ώστε να μπορέσω να καταλήξω συμπεράσματα. Πρέπει να πω ότι με ικανοποίησε πάρα πολύ ο τρόπο με τον οποίο διεξήγησαν οι συνεδρίε σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο συνεδριάσεων, όχι μόνο διότι υπήρχε μεγάλη ε, αριθμό συμμετεχόντων, 70 έως 100 άτομα θα έλεγα, αλλά επίσης με εντυπωσίασε και η ποιότητα των συζητήσεων. Όπως είπα, οι συνεδριάσεις άρχισαν στις 11 Ιανουαρίου με την παρουσίαση της ανακοίνωσης και τις υπόλοιπες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσει να ε, δοθεί μια νέα πνοή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο υπεύθυνος της ομάδας Market και η ομάδα του μας παρουσίασαν το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πράσινη βίβλο για ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής και η κυρία Μάινορ, υπεύθυνη τη ΣΑΝΚΟ για θέματα καταναλωτών, παρουσίασε τη μελέτη για την συμπεριφορά των καταναλωτών στις αγορές online ε, την ίδια μέρα. Στη δεύτερη συνεδρίαση χωρίσαμε τις ε, συζητήσεις σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα τις ε, συμβάσεις οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά και τον τρόπο τον οποίο μπορεί να γίνει ο εντοπισμός ε, κάποιων στοιχείων. Ήταν ο κύριος Αλαντεκέας παρόν, υπεύθυνο για το e-procurement, υπεύθυνο για τις ε, κρατικές προμήθειες, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος παρουσίασε σύντομα τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε σχέση με το e-procurement πολλές από τις οποίες παρουσιάστηκαν στην ε, Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου και πρόσφατα στη διάσκεψη που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες για το θέμα αυτό των ε, ηλεκτρονικών κρατικών προμηθειών. Επίσης είχαμε τις απόψεις του ιδιωτικού τομέα με τον κύριο, την παρουσίαση του κύριου Ενρίκ Μπουρντέλ, οποίος είναι εμπειρογνώμων και σύμβουλος σε θέματα τέτοιων πολιτικών. Και θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα ότι κατά την άποψή μου οι ηλεκτρονικές συμβάσεις είναι πολύ πιο σημαντικές ε, από ότι οι κλασικοί τρόποι που χρησιμοποιήσαμε, διότι έτσι όλες οι κρατικές προμήθειες και οι συμβάσεις που τις ε, ακολουθούν γίνονται πολύ πιο διαφανείς για όλα τα μέρη. Και έτσι πιο αποτελεσματικές και μπορούν να οδηγήσουν και σε αποτεμίευση κονδυλίων από τη, εκ μέρου των, της δημόσιας διοίκησης σε κάθε χώρα, πράγμα πιο αναγκαίο από ποτέ σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε πώς να εξοικονομήσουμε χρήματα των καταναλωτών, των φορολογουμένων και με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρουμε σε αυτό. Η δεύτερο πάνελ ασχολήθηκε με την ε, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική υπογραφή με τη βοήθεια του κυρίου Γκαλέρ και της κυρίας Βάιλντερ που μας μίλησαν για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα θέματα αυτά. publicados con la nueva propuesta. Και ακούσαμε και τη νέα πρόταση για την ρύθμιση του θέματος αυτό της ηλεκτρονικής υπογραφής. Είχαμε και τον κύριο Τίλμαν σύμβουλο της European Affairs του Eurochambers, την συνεδρίαση που μας μίλησε για τα πλεονεκτήματα των μέτρων αυτών για τις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολλά τα πλεονεκτήματα. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα όσον αφορά την ηλεκτρονική ε, υπογραφή και την πιστοποίηση. Ασχοληθήκαμε και με το νέο νομοθετικό πακέτο που πρότεινε η Επιτροπή για θέματα προστασίας δεδομένων. Πρόκειται για πρόταση που θα έχει μεγάλε επιπτώσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ανταλλάξαμε επιχειρήματα και απόψεις. Κυρία εισηγήτρια, η κυρία Μαριελέν Μπουλονζέ, υπεύθυνη του θέματος αυτό στην Κομισιόν για την μελέτη των μέτρων, καθώς και τον κύριο Χίκμαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εποπτείας ε, και Προστασίας Δεδομένων, καθώς και εκπροσώπους της Google, Mota, of Europe, που μαζί με διάφορους εμπειρογνώμονες μας είπαν πώς μπορούμε σε αυτό το νομοθετικό πακέτο να έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Πράγμα σημαντικό γιατί συζητήσει θα γίνει το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. Επίσης, μιλήσαμε για προβλήματα που έχουν οι λιανοπολιτές στο ε, διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Συνεισέφεραν ο κύριος Γκράχαμ Γουίν από τη Eurocommerce ο κύριος Σάντσες Δεμόθα και ο κύριος Τζον Έγγελς από το EMRH. Έγινε παρουσίαση και κάποιων μελετών που έκανε και η Boston Consulting Group και είδαμε και muestran de manera clara el enorme potencial del comercio electrónico para contribuir. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Είπαμε λοιπόν θα πρέπει τα εμπόδια που υπάρχουν στην Ευρώπη να τα ξεπεράσουμε το συνομότερο δυνατό. Επίσης παρουσιάστηκε και μία ε, σύμβαση τύπος για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο. Στην πέμπτη συνεδρίαση συνειδήσαμε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πρωταρχική σημασίας. Η ενιαία ψηφιακή αγορά και ο ρόλος των ΜΜΕ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι δυνατότητες που μας προσφέρει κυρίως για τις ΜΜΕ το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εξαιρετικές. Πολλές θέσει εργασία δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και η ψηφιακή οικονομία νομίζω ότι μπορεί να μα βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση αν πραγματικά δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον στο οποίο θα κινούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσει για να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και κυρίω για να ε, μπορέσουν να προσλάβουν νέου. Στι ΜΜΕ, οι ΜΜΕ για να μπορέσουν να προσλάβουν καμιά δεκαριά άτομα θα πρέπει να έχουν ε, την ε, εμπιστοσύνη ότι κινούνται στο κατάλληλο κλίμα. Πρώτα απ' όλα αυτό θα γίνει με απλοποίηση των συστημάτων, με εμπιστοσύνη στο σύστημα, στις εναλλακτικέ λύσεις που προσφέρονται ε, οι επιχειρήσεις για να ακολουθήσουν αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο εμπορίου, καινοτομία, μέσω των προγραμμάτων Ορίζων 2020 και Κόσμο, ο κύριος Μισελ Κατινά της Γενικής Διεύθυνσης Enterprise Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας μίλησε για τις διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ και για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές να ξεπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν και να κάνουν καλύτερη κατάρτιση των υπαλλήλων τους. Στη συνέχεια, η Αντίντα Σινεφ, από την ε, μονάδα Competition μας μίλησε για τις κύριες πρωτοβουλίε. παρούσες και προβλεπόμενες για την ενίσχυση που μπορεί να προσφέρει σε θέματα ΜΜΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Και τελικά ασχοληθήκαμε ένα θέμα μεγάλης σημασίας που είναι η προσβασιμότητα για όλους του ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως για άτομα τα οποία λόγω μίας κάποιας αδυναμίας δεν μπορούν προς το παρόν να έχουν πλήρη πρόσβαση. Θα πρέπει κυρίως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορέσουν όλοι να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την πρόσβαση στην ηλεκτρονική αγορά. Μιλήσαμε για περισσότερο από 60 εκατομμύρια άτομα που έχουν μια κάποια δυναμία, μια κάποια αναμυρία και δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ψηφιακό κόσμο. Η κυρία Μπάρμπαρα Μαρτίν και ο κύριος Εουχένιο Πέρεθ, Πετσαρμάν, από την ε, Εθνική Οργάνωση Τυφλών της Ισπανίας, την ΟΝΦΕ, συνεισέφεραν σε αυτή την συζήτηση. Επίσης, Είχαμε και την αντιπρόεδρο της Κυρίας Επιτροπής, την κυρία Νέλη Κρός και τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, τον Επίτροπο, που μας μίλησαν για τις κύριες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στις υπηρεσίες τους και για τις προσεχείς δράσεις που σκέφτονται να αναλάβουν για να μπορέσει να υπάρξει όντως η mm. πραγματοποίηση της ενιαίας εσωτερικής ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Στην τελευταία συνεδρία, στην 7 παρουσιάστηκαν οι διάφορε μελέτες που αφορούσαν το ενιαίο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι διάφορες μελέτες οι οποίες μαζί τη ΣΥΝΚΟ να κάνουμε μελέτη των δυνατοτήτων και ευκαιριών να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό εμπόριο ποιότητα για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών που έγινε από την Civic Consulting μελέτη για τα νομοθετικά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τον καθηγητή Πανεπιστημίου Όσναμπρουκ, μελέτη για τις δυνατότητες και τα εμπόδια για την απλοποίηση και τον εξυγχρονισμό του ΦΠΑ στο ενιαίο ε, ηλεκτρονικό εμπόριο που έγινε από την Copenhagen Economics, μελέτη για το cloud computing που έκανε η Civic Consulting και τελικά οι δυνατότητες ε, πρόσβασης στο ίντερνετ. Πρέπει να πω ότι οι μελέτες αυτές είναι εξαιρετικής ποιότητας. Mm. Σε κάθε μία από αυτές αναλύονται εξαιρετικά τα θέματα mm. τα οποία ασχολείται και βρίσκονται βεβαίως και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάθεσή σας. Ο κύριο Φρανκ Μποσιέρ από την Γελική Διεύθυνση Info έκανε και μία παρουσίαση για του μελλοντικού στόχους της ηλεκτρονικής agenda στην Ευρώπη και, μας, και πρέπει να πούμε ότι και η Κομισιό μας είπε ότι θα κάνει αναθεώρηση ε, της πρότασης Πρέπει να πω ότι ό,τι κάναμε ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Τα πρακτικά και τα πορίσματα θα δημοσιευθούν σε ένα έγγραφο το οποίο θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και θα έχετε στη διάθεσή σας και εσείς και όλος ο κόσμος. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα ήδη στα αγγλικά τα αποτελέσματα. Δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα που αφορούν το ενιαίο ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε τους επόμενους μήνες, όπως το νέο πακέτο για τα πνευματικά δικαιώματα, δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην υπάρχουν εμπόδια στα υπηρεσίες, επικαιροποίηση ψηφιακή ε, ψηφιακής και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να μελετήσουμε πιο διεξοδικά. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε μετά το ε, καλοκαίρι και άλλε συναντήσει η ομάδα εργασία. αν εσεί, ο πρόεδρο και οι συντονιστέ, το κρίνετε απαραίτητο για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Γι' αυτό θα ήθελα να παρουσιάσω επισήμως αυτό το αίτημα για να ανανεώσετε την εντολή που έχετε δώσει σε αυτή την ομάδα εργασίας μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές για να συνεχίσουμε την εργασία. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Well, thank you very much indeed. Ευχαριστούμε εμείς. Όπως είπαμε, οι εκδηλώσει θα είναι στα αγγλικά, αλλά θα υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες. Ήθελα να ευχαριστήσω την Τζοανάπα που βρίσκεται εδώ πάνω μαζί μου και διαχειρίζεται την όλη διαδικασία μαζί σου. Είναι πολύ μεγάλο το έργο σας. Πολλές μελέτες στις οποίες αναφερθήκατε. Είχαμε την μελέτη για το υπολογιστικό νέφος και για τα σημεία εξοπιστία για την προστασία δεδομένων. Όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα σύντομα και έτσι θα έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε στις διακοπέ μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μα για σχόλια. Δεν ξέρω αν κάποιος θα, θα ήθελε να σχολιάσει. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λαμότα από την Γενική Διεύθυνση και θα ήθελα να τον καλέσω να σχολιάσει αλλά πρώτα απ' όλα ας ακούσουμε τον ε, καθηγητά Κόρια Ντεκάμπος κάποιος άλλος θα ήθελε να σχολιάσει Άντωνη Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρο πριν από 18 μήνες αρχίσαμε αυτή τη δουλειά και στην αρχή ξέραμε πολύ λίγα πράγματα, πολύ γενικά όσον αφορά τις δυσκολίες Ξέραμε ότι το θέμα αυτό αφορούσε το ΦΠΑ, τις πιστοτικές κάρτες, ε, την ε, παράδοση ηλεκτρονικών προϊόντων, ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ξέραμε ότι υπήρχαν προβλήματα στον τομέα αυτό, που ήταν διακρίσεις σε σχέση με την υπηκότητα, εάν έκανε κανείς ηλεκτρονικές αγορές, το θέμα της γλώσσας, όλα ήταν στα αγγλικά, προβλήματα με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, θέματα ασφάλειας όσον αφορά τις διάφορες ιστοσελίδες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, γενικά πράγματα. Και 18 μήνες μετά πρέπει να πω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε γνώσεις γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν ε, στον τομέα αυτό. Ο Παύλο Άριες έκανε διεξοδικά την παρουσίαση των συμπερασμάτων στο οποίο καταλήξαμε, έθιξε πολλά θέματα, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, προστασία δεδομένων, στάνταρ ηλεκτρονικές συμβάσεις, ΜΜΕ και πάρα πολλοί εμείς ε, οι βουλευτές ακούσαμε τους εκπροσώπους της Κομισιόν, τους ενδιαμπλεκόμενους ενδιαφέρομενους φορείς, τους επιτρόπους, οι επιτρόπους όπως ελέγχθη κάποια φορά και έχουν εμπλουτιστεί γνώσεις μας σήμερα. Είμαστε λοιπόν σε θέση να πούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι σκεφτήκαμε στην αρχή. Γιατί το λέω, γιατί τώρα ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρως την εργασία που επιτελέστηκε και θα ήθελα και εγώ να υπεστηρίξω την ιδέα η ομάδα αυτή εργασίες να συνεχίσει τις ε, συναντήσεις και τις εργασίες της μετά από τις καλοκαιρινές δικοπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ ενθαρρυντική υποστήριξή σα. Ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα αυτό. Πρέπει να κανονίσουμε ο κύριο Άρια να έρθει να μιλήσει στου συντονιστέ ε, με μια συνοπτική παρουσίαση των επόμενων θέματων που θα καλυφθούν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το Σεπτέμβριο για να προγραμματίσουμε την επόμενη φάση των εργασιών και ενδεχομένω να το συνδέσουμε αυτό με την ατζέντα μα για τον επόμενο κύκλο εργασιών μετά το 2014. Θα μπορούσαμε να μα βοηθήσει και η Κομισιόν ενδεχομένω άλλα μέλη που θα ήθελαν να σχολιάσουν. Κυρία Λαμότ, θα θέλατε να κάνετε κάποια σχόλια εκ μέρου τη Γενική Διεύθυνση Αγορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια. Η Κομισιόν θα ήθελε να ευχαριστήσει την ΙΜΚΟ και ειδικότερα τον κύριο Παύλο Αρίας Σεβερία για την οργάνωση των συνεδριασιών του που αποτέλεσαν αναπόφευκτο σημείο συνάντηση ώστε να προχωρήσουμε στους διάφορους φακέλους αυτού του πολύπλοκου θέματος. Ε, διάφοροι φάκελοι έχουν διάφορες πτυχές. Επίσης, ε, και εμεί θα είμαστε ικανοποιημένοι αν συνεχίσει ο κύκλο συνεδριάσεων όταν γυρίσουμε από τι διακοπέ. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ουσιαστικά δεν έχουν περάσει ακόμα ούτε καν οι πρώτοι έξι μήνε ενό σχεδίου δράση ε, τετραετού ε, ή τεσσεράμιση χρόνων. Συνεπώ, αναμένουμε τη συζήτηση με όλου του εταίρου για του διαφορού φακέλου. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much. And, um... Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω λοιπόν ότι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Όλοι θα έχουν μια ευκαιρία να δουν τη σύνοψη των εκθέσεων που συνιστώ να κοιτάξετε, να δείτε τη μεγάλη γκάμα σημείων που καλύπτονται και θα καλέσουμε τον κύριο Αρίας πιστεύω, και τα άλλα μέλη των διαφορών ομάδων να προετοιμάσουν μια σύνοψη για τις εργασίες του επόμενου εξαμήνου για αυτή την ομάδα και να σχετιστεί με τις προτάσεις που εξετάζουμε. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν εξαιρετικά. Επίσης, καλό θα ήταν να έρθουμε σε επαφή με άλλες επιτροπές που εμπλέκονται επίσης. Υπάρχουν πολλές άλλες επιτροπές ουσιαστικά που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Και η κυρία Κρέμη φυσικά θα έχει ρόλο κλειδί όσον αφορά την οδηγία προστασίας δεδομένων η γνωμοδότησή μας για αυτή θα είναι εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο των εργασιών μας μέσα στο επόμενο εξάμενο και πέραν αυτού. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για όλα αυτά. Είναι 10 η ώρα και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην ημερήσια διάταξη που έχουμε μπροστά μας. Η κυρία Γκαλπέλτσο είναι εδώ πίσω από την κάμερα. Ε, σας πειράζει να μετακινηθείτε διότι χρειάζομαι να βλέπω την κυρία Γκάλπελ. Ε, σηκώνει το χέρι της. Ε, έχουμε μια ταινία για την ψηφοφορία ADR. Ε, γι' αυτό βρίσκεται εδώ ο κάμεραμαν, αλλά μπορείτε να έρθετε αργότερα, κύριε Γκάλπελ. Πρέπει να φύγει να παρεψηφίσει μια άλλη επιτροπή. Ε, έχει ελάχιστε τροπολογίε για τη γνωμοδότησή τη σε σχέση με τι 700 που υπάρχουν για τι επόμενε. Ε, Σα πειράζει να πάρουμε πρώτα τη δική τη, να εξετάσουμε πρώτα τη δική τη ε, γνωμοδότηση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει πρώτα να μελετήσουμε τη γνωμοδότηση, να ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση της κυρίας Γκάλ Είναι όλοι έτοιμοι να ψηφίσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε απαρτία, αλλά Μπορώ να έχω την προσοχή σας λοιπόν. Κύριε Γκαλπέλτς, θέλετε να πείτε κάτι πριν προχωρήσουμε στη ψηφοφορία για την εκθεσή σας. Όχι. Ωραία. Χρειαζόμαι λοιπόν την λίστα ψηφοφορία για αυτά. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για την γνωμοδότηση της κυρίας Γκάλπελτς. Είστε όλοι έτοιμοι. Ωραία. Η κυρία Ρούλε απέσυρε την τροπολογία της για απόρριψη. Θέτω λοιπόν στην ψηφοφορία την τροπολογία 1 του, της συγγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 του κυρίου Ντε ηλεκτρονική ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία ώστε να ελέγξουμε και τη λειτουργία του συστήματος. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την τροπολογία 39 του κ. Ιόγκ. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, 27 έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμή. Από 32 δεν ξέρω αν θέλει να ψηφίσει και κάποιο άλλο. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για τη συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάω τώρα στην τροπολογία 2 της ηγετρίας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 4 της ηγετρίας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 του κ. Ντεγιόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 50. Υπάρχει ένας επιπλέον σοσιαλιστής, ε, θα, μπορούσε, θα πρέπει κάποιος να βγάλει την κάρτα του. Βγάλετε μια κάρτα, σοσιαλιστές. Κυρία Πέντεργαστ, ευχαριστώ. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51 της κυρίας Παρβανόβα και Γκαλπέλ, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 53 του κυρίου Μάντερ υπέρ, κατά, Εποχές εγκρίνεται 52 του κυρίου Ντεγιόγκ άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Μια ψήφος κάνει μια μεγάλη διαφορά. 54 του κ. Μάντερς υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 η, της κυρίας Γκαλπέλτσο υπέρ κατά 5 συγγνώμη υπέρ κατά εγκρίνεται 6 και 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 της συγκήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 57 του κυρίου De υπέρ άρχεται η ψηφοφορία συγγνώμη για την 57 εξακολουθούμε να έχουμε ένα μέλος των σοσιαλιστών παραπάνω. Είμαστε 11 λέει κυρία Πέντρεγκαστ. Αλλά σύμφωνα με το μηχάνημα έχουμε ένα παραπάνω. Κάποιος λοιπόν Για ελέγξτε το. Εδώ είμαστε 11. 11. Να ακυρώσουμε αυτή την ψηφοφορία. Μπορούν τα μέλη των σοσιαλιστών να ψηφίσουν τώρα όλα τα μέλη παρακαλώ. Μπορείτε όλοι οι σοσιαλιστές να ελέγξετε και να ψηφίσετε όλοι αυτή τη στιγμή μόνο σοσιαλιστές. Σοσιαλδημοκράτες. Ωραία, σωστά λοιπόν. Θα επαναλάβουμε τώρα την ψηφοφόρια. Λοιπόν, υπήρχε σαφώς ένα άτομο παραπάνω. Ε, η οθόνη τώρα μέτρησε 11 μέλη. Νομίζω ότι ψήφιζε κάποιο άλλο, αλλά δεν πειράζει τώρα. Το κυρώσαμε. Α επιστρέψουμε τώρα στην τροπολογία 57 του κυρίου Ντέγιονγκ, Άρχεται η ψηφοφορία. 34 κάρτες υπάρχουν μέσα, αλλά 30 ψήφισαν μόνο. Κάντε γρήγορα, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 58 και 59 τροπολογίες του κ. Ντεγιόν και της κ. Αλδεμόσα. Άρχεται η ψηφοφορία για τις 58 και 59. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται επίσης. 60 του κ. Ντεγιόγκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται επίσης. Τροπολογία 8 την Καλπέλτσο υπέρ κατά αποχές εγκρινέται 61 του κυρίου Ντεγιόγκ. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία για την 61. Να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ γιατί τελειώς θα περάσουμε όλη την ημέρα. Εδώ κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 62 του κυρίου Ντεγιόγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 του κυρίου Μπίλαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 64 καταπίπτει λοιπόν 65 η, του κυρίου Μπίλαν υπέρ κατά απορρίπτεται καθαρά 66 του κ. Ντεγιόγκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 του κ. Ντεγιόγκ εξεκινάει ψηφοφορία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 Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 21. Είναι συμβατή. Μπορούμε να την ψηφίσουμε υπέρ της 21. Δεν χρειάζεται λέει, να ψηφίσετε για την 21. Η 21 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Επειδή ε, εγκρίναμε την 73. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 79 υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία. Κλείνει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Η... Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 25. Κλείνει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε μαζικά τις τροπολογίες του κύριου Ντεγιόγκ. Ναι, όχι. Ωραία, ας τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Περνάμε λοιπόν στην 26. Θα τις δούμε ξεχωριστά. 26 ε, ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μπορούμε ίσως να το κάνουμε και με ανατασχέων. ...27 ε, απορρίπτεται, 28 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται, 29 υπέρ, 29 υπέρ. Να ψηφίσουμε. 29. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 29. Δύο πλειοψηφίε διαφέρουν. Γι' αυτό κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 31 από την κυρία Σόλδεμο. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 32 με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 36 ξεκινάει η ψηφοφορία για την 36 ηλεκτρονικά κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται κατά δύο ψήφους 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα θα έχουμε την όλη γνωμοδότηση στη ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία Ξεκινάει η ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης. Uh, ε, is... Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 36 ψήφοι υπέρ, καμία κατά. Ευχαριστούμε κυρία Γκαλπέλτσε. Αυτό... Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υπερασπίσετε τη θέση μας στην Επιτροπή Μεταφορών ή σε οποιαδήποτε Επιτροπή ασχοληθεί με αυτό. Ναι, Επιτροπή Μεταφορών. Ε, Τώρα η έκθεση του κ. Κορέ. Για να δω στον κατάλογο ψηφοφορίας μήπως θέλει ο συγητής να μας πει τίποτε προκαταρκτικά. Όχι, εντάξει. Πάμε. Η κάμερα είναι από την ε, εσωτερική μας υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, που κάνει ένα ρεπορτάζ. Article 1, compromise amendment. Λοιπόν, συμβιβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 227 του κυρίου Φόξ. Άρχεται η ψηφοφορία. Μλήξε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Περ. Κατά. Εγκρίνεται. 233. Ηλεκτρονικά. Σας παρακαλώ ψηφίζετε γρηγορότερα, δεν θα προλάβουμε. Έληξε. Εγκρίνεται και αυτή. 234 υπέρ. Α, πάλι επαλήθευση για την 234. Αλλά παρακαλώ να πατάτε τα κομπιά γρήγορα γρήγορα. Τσαμπούκ, τσαμπούκ. Έλξε. Εγκρίνεται και αυτή. 47 και άλλες υπέρ κατά α μια στιγμή μια στιγμή, μια στιγμή. Φόξ και άλλων λοιπόν ε, πάλι, όχι ε, με τα χέρια ξανά υπέρ κατά «47 Γκρέκ 235 Φόξ και νομικής 21». Αυτά ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ λοιπόν. Α, όχι, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Κα. Έλξε. Εγκρίνονται. 236 έχει αποσυρθεί. 237 φόκτ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 242 Fox δύο τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 244 Σαλτεμόζε ηλεκτρονικά έληξε εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 καλύπτεται από τη συμβαστική. 57 υπέρ κατά εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 261 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 262 καταπίπτει, 263 ηλεκτρονικά. έληξε είπα 263 έληξε εγκρίνεται άρα καταπίπτει 59 συμβιβαστική 9 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 323 έχει αποσυρθεί 62 έχει αποσυρθεί 63 τι υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται η 267-268 καταπίπτουν και 269 καλύπτεται από το συμβιβασμό και 39 νομικής όχι 268 πιάστηκα 268 ως προσθήκη αφού εγκρίθηκε η 63 λοιπόν ηλεκτρονικά για την 268 έληξε εγκρίνεται ως προσθήκη νομικής 40 Α, ε, ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά νομική 40 ηλεκτρονικά έληξε εγκρίνεται 274 Fox υπέρ κατά Απορρίπτεται. Νομικής 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομικής 26 δεν την ψηφίζουμε γιατί καλύφθηκε καθώς και πολλές από τις υπόλοιπες. Συμβιβαστική 10. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Ποιε εγκρίνεται. Νομικής 28. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 66 του εισηγητή υπέρ. Όχι, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Μλήξε. Καταπίπτει, δηλαδή απορρίπτεται. Με ψηφία. 2.94 ποπάκι. Ηλεκτρονικά. έληξε απορρίπτεται 295 υπέρ κατά απορρίπτεται 67 υπέρ κατά εγκρίνεται 296 και νομικής 29 ηλεκτρονικά έληξε εγκρίνεται 68 του συγητή. Ο 297 έκανα λάθος του συγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 298 του κυρίου Μπουσόη για να προσθεθεί η λέξη όπου χρειάζεται. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ πατάτε τα κουμπιά πιο γρήγορα σας το ξαναείπα και πριν. Λίγη. Εγκρίνεται. 299 και νομικής 30 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 68 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται καταπίπτει 300. Επομένως νομικής 31 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 70 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Νομικής 32 έχει καλυφθεί 301 φόξ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 71 υπέρ, 71 υπέρ δεν είναι σαφές, 71 ηλεκτρονικός έληξε ισοψηφία απορρίπτεται. Άρα καταπίπτει και η 302. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Νομικής 33. Νομικής 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. 72 ηλεκτρονικά. 72. Ξέρει. Εγκρίνεται. 302 με μία προσθήκη with due regard for data protection. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 303 επομένως καταπίπτει, 73 υπέρ κατά εγκρίνεται. 304 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 305 και νομικής 34. Υπέρ. Όχι. Ηλεκτρονικά. 305 Μπουσόη. Θέλατε να πείτε τίποτα κύριε Μπουσόη. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν σε όλες τις μεταφράσεις τη σωστή έκφραση. Δεν λέει όπου χρειάζεται, αλλά όπου υπάρχει. Όχι στείλα λαπλή αλλά if available. Ευχαριστώ. Α, δηλαδή η προσθήκη είναι όποτε υπάρχει. Μάλιστα. Ψηφίζουμε. Είστε υπέρ, ε, μάλιστα. Υπέρ. Όχι, πρέπει ξανά ηλεκτρονικά. Άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 74 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 306 πίπτη. 75 και νομική 35 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 307 πίπτη. 76 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. νομική 36 υπέρ. Κατά. Δεν συγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Νομική 37 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 313 κατά πίπτη. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 320 κατά πίπτη για την κρίση του συμβιβασμός. 321 που πάκι ηλεκτρονικά. Έλξε απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά εγκρίνεται 324 κατά τη νομικής 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 80 υπέρ 80 υπέρ κατά εγκρίνεται νομικής 42 δεν την ψηφίζουμε 325 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται 326 έχει αποσυρθεί 81 υπέρ κατά εγκρίνεται 82 υπέρ κατά εγκρίνεται ή 328 κατά πίπτη 329 επίσης 83 υπέρ όχι ηλεκτρονικά έληξε απορρίπτεται με ισοψηφία. τέλο πάντων, έχουν λίγο κάποιο μπέρδεμα εδώ γιατί ψηφίζουν μάλλον περισσότεροι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η 333 καταπίπτει. Μα απορρίφθηκε η 83. τότε θα ψηφίσουμε την 333. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 330 ως προσθήκη στην 333. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 331 και 332 αλλά την 84 υπέρ. Κατά. Ποιες συγκρίνεται. 334 και 336 κατά πίπτουν και οι 335 νομική 45 υπέρ κατά ποιες συγκρίνεται 85 υπέρ κατά ποιες συγκρίνεται οι 337 και 338 καταπίπτουν 339, 340 έχει αποσυρθεί 342 υπέρ ηλεκτρονικά. Έληξε. Απορρίπτεται από την ισοψηφία. 18-18. 341 υπέρ κατά εγκρίνεται 86 κατά καταπίπτει 343 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 87. Ο συμπληρωματική. Υπέρ. Κατά. Ε, έλεγχος. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3.44 καταπίπτει. 3.45 αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 3.46. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 3.47. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 3.48. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 3.49 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3.50. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 88 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 351. Φόξ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, 44. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων 355 και Τζούρι 48 47 με συγχωρείτε απορρίπτονται 91 υπέρ κατά συμβιβαστική 15 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 16 υπέρ κατά εγκρίνεται νομικών υποθέσεων 51. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 372 καταπίπτει. 96. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 373 υπέρ κατά εγκρίνεται. Καταπίπτει 374, 375 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά απορρίπτεται. 376 καταπίπτει. Όχι. Όχι. Την ψηφίζουμε. 3,76. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3,78. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τζούρι 52. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3,79 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 98, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. «136. Υπέρ κατά εγκρίνεται». 102 υπέρ κατά εγκρίνεται 103 εγκρίνεται Τζούρι 54 με προφορική τροπολογία Μπουσόη. Είστε υπέρ της αλλαγής της διατύπωσης. Έχει καλώς. Ε, με την αλλαγή που έγινε προηγουμένως τη λέξη available. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 387. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τζούρι 55 ως προστίκι Υπέρ κατά εγκρίνεται. The vote's closed. That's carried by one vote. Um, so 107 falls. 389. 389, uh, the vote is open on 389. Uh, the vote is closed. Η 20 σελίδα αυτού νου λείπει. Δεν πειράζει. Uh, so 108 falls. 390. Καλύπτεται η 390 από τη συμβαστική. 109 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τον 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τζούρι 56 ως συμβιβαστική. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά εγκρίνεται. 391 de Jong απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά εγκρίνεται. Καταπίπτει 57 της Τζούρι, 114 υπέρ κατά εγκρίνεται. Καταπίπτει Καταπίπτουν οι 58, 392 και 393, 394 Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Και πάλι θέλω να ξαναψηφίσετε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 395 και καταπίπτει ως προσθήκη 59 της Τζούρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 120. Υπέρ κατά εγκρίνεται 121 υπέρ κατά εγκρίνεται 122 υπέρ κατά εγκρίνεται 397 υπέρ κατά απορρίπτεται 396 υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική ψηφοφορία Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψήφο. Χωριστή ψηφοφορία που ζήτησε η Άλντε για την 398. Το ε, πρώτο μέρος αφορά την αλλαγή από 18 σε 24 μήνες. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος Το δεύτερο μέρος αφορά όχι πρόσθεση, αλλά διαγραφή. Υπέρ. Κατά. That's clearly rejected. Yeah. That was clearly rejected. Yeah. So, so the words stay. That's yeah. yeah. So there's no change to Rule 398. Um, and so... Τι γίνεται με το 399. Έχουμε δύο φορές. Well, none of it's been adopted. No. Well, we didn't adopt either the first or the second part of 399. All right. Can we vote on 399? All right. We can vote on 399. So 399, uh, 399, the vote's open on 399. 99, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο υπέρ περισσότερη. 401 υπέρ κατά απορρίπτεται. 400 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 123. 402. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 126 υπέρ. Εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ. Πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι. Τροπολογία αριθμός 1. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παρακαλώ, για να πηγαίνουμε γρήγορα, σηκώστε το χέρι όταν χρειάζεται έγκαιρα. Δύο ηλεκτρονική επαλήθευση. η φιλελεύθερη παρακαλώ τα χεράκια. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επαλήθευση αν οι φιλελεύθεροι υπερψήφισαν. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θέλει κανεί να κάνουμε ηλεκτρονική πελίδευση. Όχι. Καταπίπτει 128 σε αυτή την περίπτωση. Καλύπτεται 129 από την 4 και περνούμε στην 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 131, η Τζούρι 1, η 130 Και τώρα πηγαίνουμε στην τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Καταπίπτει 133, 8, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τζούρι 2, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 9, υπέρ, κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά απορρίπτονται 11 Φιλελεύθερη παρακαλώ. Those in favor, please. Υπέρ παρακαλώ. Υπέρ της 11. Κατά. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 135. Υπέρ. Εδώ χρειαζόμαστε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Εντάξει. Απορρίπτεται. Δεκατρεις. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τζούρι 3 ως προστίκη, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η αιτιολογική σκέψη θα καλύπτεται από την ε, συμβιβαστική. 143 ζουβά υπέρ κατά απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Προσπάθησα να πάω πιο γρήγορα, αλλά... Λοιπόν, 144 ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Το, οι 11 και οι 12 καλύπτουν τη συμβαστική 6 και 3. Πάω στη τζούρι 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 152. 154. 100. 53 καλύπτω τις 158 γκρέχ. Η 157 ως προσθήκη. Συμβιβαστική 19. Υπέρ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 160. Υπέρ. 160. Θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ξεκλίνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Τώρα ψηφίζουμε για την 161. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 19. Καταπίπτει συμβιβαστική 20. Συγγνώμη. Τροπολογία 19 ως προσθήκη. Υπέρ. κατά 19 υπέρ κατά η φρέλευθερη πάλι δεν ήταν βέβαιη τροπολογία 19 λοιπόν οι αναποφάσιστοι δεν είναι σίγουροι προ, ποιος, προς ποια πλευρά δεν αποφασίζουν ψηφίστε λοιπόν παρακαλώ πιο γρήγορα κλείνει η ψηφοφορία Εγκρίνεται. Κατά πέντε ψήφους. Οι φιλελεύθεροι όμως ψήφισαν υπέρ. Ωραία, λοιπόν. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 21 του κ. Γκρέχη υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Ξεκινάμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 22. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται κατά μία ψήφο. Τροπολογία 163 καταπίπτει και περνάμε στην νομικών υποθέσεων 7. Όλες αυτές καλύπτονται από τις συμβαστικές. Περνάμε λοιπόν στην 169 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται η τηλεογική σκέψη 19 καλύπτεται από τη συμβιβαστική 12 ε, έχουμε λοιπόν την 174 ε, ξεκινάει η ψηφοφορία για την 174 τροπολογία κλείνει η ψηφοφορία Απορρίπτεται. Η αιτιολογική σκέψη 20 καλύπτει από τη συμβιβαστική 11, 21, συγγνώμη, λάθος, 181 του εισηγητή για την αιτιολογική σκέψη 21. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 28, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 και 14 έχουν καλυφθεί. Περνάμε στην τροπολογία 193 και Γιούρι 14. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τις 193 και Γιούρι 14. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται κατά μία ψήφο. Συμβιβαστική 11 καλύπτει την επόμενη ομάδα τροπολογιών. Περνάμε λοιπόν στην 33 και 186 που είναι ίδιες. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τις, για τις 33 και 186. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορριπτούνται. Τροπολογία 185. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 187 και 91 αποσύρονται. Η αιτιολογική σκέψη 22 καλύπτεται από τη συμβιβαστική 16. Περνάμε στην τροπολογία 35, προφορική τροπολογία της, του εισηγητή. Διαγραφή, το βλέπετε εδώ, ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 196 καταπίπτει, 198 αποσύρεται. Περνάμε στι νομικέ υποθέσει 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. 197 ως προσθήκη στην γιούρη 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται Συμβαστική 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 39 Κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται κατά δύο ψήφους. 199 έως 201 καλύπτονται αυτή 39 202 λοιπόν υπέρ πρέπει να το θέσουμε σε ψηφοφορία ξεκινάει η ψηφοφορία για την 202 κλείνει απορρίπτεται κατά μία ψήφο νομικές υποθέσεις 11 καλύπτεται από τους συμβιβαστικές περνάμε τροπολογία 203 υπέρ ξεκινάει η ψηφοφορία για την 203 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται κατά δύο ψήφους 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά 205 υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς ε, τροπολογία 40 και 208 υπέρ κατά εγκρίνεται 207 καλύπτεται και 206 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 41 με ψηφοφορία κατά τμήματα που ζήτησε η Γκουε. Ας πάρουμε το πρώτο κομμάτι. Πρώτο κομμάτι 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με την προσθήκη των λέξεων αυτών του κειμένου αυτού. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία γι' αυτό. Κλείνει ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά τρεις ψήφους. 210, 211 και γύρω 17 καταπίπτουν όλες. Περνάμε στη 213 του κύριου Γκρέχ. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 42, 43. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 145 καταπίπτει 215 υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς 214 ξεκινάει η ψηφοφορία για την 214 κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται κατά μία ψήφου 216 υπέρ κατά εγκρίνεται Ε, τα citations 1, 2... Η αιτιολογική σκέψη 1 και 2. Ευχαριστούμε πολύ. Τελική ψηφοφορία. Σας ευχαριστούσα απλά για την πολύ αποτελεσματική ψηφοφορία σε ένα τόσο μεγάλο θέμα ξεκινάει η ψηφοφορία για την πρόταση για την ηλεκτρονική υπηρεσία διαφορών του κ. Γκρέχ. Περιμένω να ψηφίσουν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 34 υπέρ και μία κατά. Ευχαριστούμε πολύ τον Λουί Γκρέχ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το φάκελο εξαιρετικά και όλους όσους τον βοήθησαν. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Φουντούν για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφόρων. Θέλει η κυρία εισηγήτρια να πει κάτι. Ευχαριστώ. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ανθρώπων και πολλών οργανισμών μαζί Χαίρομαι ιδιαίτερα για την περαιτέρω εργασία που θα κάνουμε με την Κυπριακή Προεδρία. Συχνά όλοι μιλάμε για την έλλειψη ατόμων που δραστηριοποιούνται online και ιδίως δυσυνοριακά με αυτή τη γνωμοδότηση θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτή την κατάσταση και θα υποφεληθεί ιδιαίτερα η εσωτερική αγορά. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για την υποστήριξή σας. Α περάσουμε λοιπόν στην εκθέση της κυρίας Τούν. Ας περάσουμε τον τίτλο. Ε, Γιούρι 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 127 του κ. Τριανταφυλλίδη υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 130-131 ξεκινάει η ψηφοφορία για αυτές τις τροπολογίες ηλεκτρονικά. Μπορείτε παρακαλώ να κάνετε πιο γρήγορα γιατί μόνο 31 ψηφίζουν τώρα. 32-33 ε, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Να σας ζητήσω, σας παρακαλώ να ψηφίζετε πιο γρήγορα, πιο ζωηρά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα. Περνάω στην Τζούρι. Τζούρι 21. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά απορρίπτεται 17 υπέρ κατά εγκρίνεται 135 αποσύρθηκε 134 υπέρ κατά απορρίπτεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 23 καταπίπτει, της Τζούρι 19 και οι άλλες παρόμοιες ε, τροπολογίες υπέρ κατά εγκρίνεται. 137 καταπίπτει, 138 υπέρ κατά απορρίπτεται, 139 υπέρ κατά εγκρίνεται, 140 και 25 γιούρι υπέρ κατά απορρίπτονται, 141 υπέρ κατά απορρίπτονται 142 και γιούρι 26 υπέρ κατά απορρίπτεται 143 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά απορρίπτεται εγκρίνεται 146 υπέρ κατά απορρίπτεται 147 υπέρ κατά εγκρίνεται Γιούρι 27 καταπίπτει, 148 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 149 και 151 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Γιούρι 29 καταπίπτει, 152 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά εγκρίνεται 155 υπέρ κατά εγκρίνεται 156 και 159 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 και 157 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται 158 υπέρ ξεκινάει η ψηφοφορία για την 158 απορρίπτεται νομίζω κατά μία ψήφο 160 υπέρ κατά εγκρίνεται 161 καταπίπτει η Γιούρι 28 υπέρ Γιούρι 28 ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση περνάμε τώρα στην Γιούρι 30. Νομικών υποθέσεων 30. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, γκρίνεται. Ε, νομικών υποθέσεων 31 υπερκατά εγκρίνεται η τζούρι 32 Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τζούρι 32 κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται κατά δύο ψήφους τζούρι 33 υπέρ κατά εγκρίνεται τζούρι 34 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται περνάμε στην 165 τώρα υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 166 υπέρ κατά εγκρίνεται 168 υπέρ κατά εγκρίνεται 169 και 170 υπέρ κατά εγκρίνεται 171 υπέρ κατά εγκρίνεται 172 υπέρ κατά εγκρίνεται 173 υπέρ κατά εγκρίνεται Η 178 καταπίπτει, 174 υπέρ κατά εγκρίνεται. 29 αποσύρεται, 179. Συγγνώμη, 175. 175 τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην 181 υπέρ ...181. Την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την 182 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 183 Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μάλλον, κατά νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 183. Εγκρίνεται. Και η γιουρή 37 κατά πίπτη συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 36 αποσύρεται 187 υπέρ κατά εγκρίνεται 188 υπέρ κατά απορρίπτεται 189 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 190 καταπίπτει Τζούρι 38 υπέρ κατά εγκρίνεται Τζούρι 39 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 39 καταπίπτει. 191 τροπολογία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 191. Ξεκινάει. Ολοκλήρωση ψηφοφορία εγκρίνεται κατά μία ψήφο. 193 καταπίπτει. 192 τι θέτουμε σε ψηφοφορία υπέρ 192 νομίζω ότι χρειάζεται να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 192. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά μία ψήφου. Τώρα περνάμε στο αρθρό 8. Έχουμε μαζικές ψηφοφορίες εδώ. Μπλοκ 1. Υπέρ για την 1. Ε, κατά εγκρίνεται. Σαφώς σημαίνει αυτό ότι οι 2 και οι 3 καταπίπτουν. Το ίδιο και οι 204-41 και περνάμε κατευθείαν στο άρθρο 8 παραγραφός 3 μαζική ψηφοφορία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο καταπίπτει και περνάμε στις 2.32, 2.33. Α, όχι, καταπίπτουν και αυτέ. Περνάμε τώρα άρθρο 8, παράγραφος 4. Περνάμε στην τροπολογία 2.45 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ψήφισμα για τη 2.46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 248 υπέρ κατά απορρίπτεται Επίση 53 υπέρ κατά εγκρίνεται 249 υπέρ κατά απορρίπτεται 54 υπέρ κατά εγκρίνεται 250 υπέρ Νομίζω ότι χρειάζεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία γιατί 2.50. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο 2.51. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά εγκρίνεται 60 υπέρ κατά εγκρίνεται και 256 και 61 υπέρ κατά εγκρίνονται 62 υπέρ κατά εγκρίνεται 63 υπέρ κατά εγκρίνεται 64 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 66 τώρα υπέρ κατά Επίση εγκρίνεται 67 υπέρ κατά εγκρίνεται 68 υπέρ κατά εγκρίνεται 258 τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται Γιούρι 57 Τζούρι 57 ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Τζούρι 57 κλείνει η ψηφοφορία Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 259 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τζούρι 58. Υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Τζούρι 58. Κλείνει η ψηφοφορία για την Τζούρι 58. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 261. Υπέρ. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. 261. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 263. Υπέρ. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 263. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 264. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς 265. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τζουρί 59. Υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά εγκρίνεται τζούρι 60 και τροπολογία 75 μάλλον ε, υπέρ κατά εγκρίνεται τζούρι 61 κατά πίπτη. τζούρι 62 υπέρ κατά ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Ξεκινάει η ψηφοφορία για την Τζούρι 62. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 266 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τζούρι 63 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τζούρι 64. Τζούρι 64. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την Τζούρι 64. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στα προαρτήματα τώρα. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά εγκρίνεται 79 υπέρ κατά εγκρίνεται 269 κατά πίτι 270 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 80 υπέρ κατά εγκρίνεται μπορούμε να ψήσουμε μαζικά για όλες αυτές ε, τις επόμενες δεν έχει κανείς αντίρρηση από την λοιπόν θα ψηφίσουμε από την 81, 82, 83, 84, 85, 86 και 87. Έχει κανείς αντίρρηση? Υπέρ. Κατά. Όλες εγκρίνονται. Περνάμε στα εκτιμώντας ε, στις επιλογικές σκέψεις. Επιλογική σκέψη 2, τροπολογία 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές επίσης απορρίπτεται τζούρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά εγκρίνεται 91 υπέρ κατά εγκρίνεται 92 υπέρ κατά 92 νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Ξεκινάει η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. 93. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Jury 3. Καταπίπτει. Τροπολογία 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τζούρι 4 υπέρ. Τζούρι 4 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τζούρι 5 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τρο... Συμβαστική 9 υπέρ. Τζούρι 2 εγκρίθηκε. Τζούρι 2 δεν ε, εγκρίθηκε. Θα την ψηφοφορία τη συμβαστική 9 εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 101 υπέρ. Κατά Δεν είναι πολύ σαφές. 101 ξεκινάμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Όταν λέει λοιπόν jury 6 ότι καταπίπτει αν εγκριθεί οποιοδήποτε από το παραπάνω Περνάμε στην τροπολογία 102 λοιπόν γιατί την η τζουρί 6. Υπέρ για την τροπολογία 102 κατά. Απορρίπτεται. Τζουρί 7. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τζουρί 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 103, 104, 105 υπέρ κατά δεν είναι πολύ σαφές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά 103 μέχρι 105. Βέβαια, και τα χέρια σας. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο. έχουμε ψηφίσει όλοι. Ναι, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 106. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10 συμβιβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται τζούρι 9 και τζούρι 10 καταπίπτουν συμβιβαστική 11 υπέρ κατά εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 112 υπέρ κατά εγκρίνεται τζούρι 11 υπέρ τζούρι 11 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Τζούρι 11. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Και εδώ νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 113. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, ξεκινάει η ψηφοφορία, κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται κατά πέντε ψήφους. 115, Τι θέτουμε σε ψηφοφορία ηλεκτρονική, α, ε, με τα χέρια, ε, υπέρ κατά, εγκρίνεται, 114 υπέρ και παρεμφερείς εγκρίνονται, τζούρι 12 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, ε, μάλλον να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ας το ελέγξουμε, λοιπόν, τζούρι 12. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τζουρί 13. Καταπίπτει. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 9 καταπίπτει, 110, είχε αποσυρθεί, συγγνώμη, 119 υπέρ κατά εγκρίνεται, 120 υπέρ κατά κοντινό το αποτέλεσμα, οπότε ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Ήταν πολύ κοντινό το αποτέλεσμα. Καταπίπτει λοιπόν. Τζούρι 14. Υπέρ κατά. Απορρίπτεται τζούρι 15. Η 68 είχε εγκριθεί, συνεπώ η Τζόρι 15 καταπίπτει. Τροπολογία 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 122 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 122. The closed. Uh, and I changed. All oh, right, that was clearly εγκρέθηκε... 123. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 123 ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. 124 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τζούρι 16 υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται 125 υπέρ κατά εγκρίνεται τζούρι 17 καταπίπτει και τζούρι 18 καταπίπτει τελική ψηφοφορία λοιπόν. α, ε, τροπολογία 12 υπέρ κατά εγκρίνεται συνεπώς τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει η ψηφοφορία για ολόκληρη την πρόταση κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ μία κατά ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστώ την κυρία Τούν και όλους τους κύριους συζητητές. Δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε πάρα πολλές γνωμοδοτήσεις ακόμη να ψηφίσουμε. Αρχίζουμε την κυρία Πετικάιναν. Παρακαλώ, όποιοι δεν θέλουν να μείνουν για τις υπόλοιπες ψηφοφορίες, να φύγουν ήρεμα από την αίθουσα. Η κυρία Πετικάινεν δεν θέλει να πει τίποτε και αρχίζουμε την ψηφοφορία της νομοδότης κυρίας Πετικάινεν. Πετικάινεν. Παρακαλώ. Προσοχή. Για να αρχίσουμε. Ησυχία παρακαλώ για την επόμενη ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Γκρέσ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2. Συμβατεί με την 1. Ε, Εγκρίνεται. Τρία. Γκρέσ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Χωριστή πληροφορία ζήτησε η ΓΟΕ. Η πρώτη χωρίς τις λέξεις υψηλό επίπεδο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το πρώτο μέρος της συμβαστικής τροπολογίας 1. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Σε αυτή την περίπτωση Λοιπόν, απορρίπτεται η συμβαστική τροπολογία. Α, να το αποσαφηνίσουμε. Ας ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα τη συμβιβαστική τροπολογία. Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, διότι νομίζω ότι στον κατάλογο υπήρχε κάποιο σφάλμα. Ευχαριστώ. Μία διευκρίνηση για όλους. Μέρος της συμβιβαστικής τροπολογίας ήταν να προσθέσουμε a high level of στο κείμενο. Πρόταση των σοσιαλδημοκρατών. Το high level of. Και μετά η Γκουε ζήτησε την διαγραφή αυτών των λέξεων. Άρα περί αυτών των λέξεων πρόκειται τώρα. The, first vote was then, uh, Άρα την πρώτη φορά ψηφίσαμε για το αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε τους όρους high level off ή όχι. Ο πρόεδρος. Ακούστε. Ας ψηφίσουμε όλη τη συμβαστική τροπολογία χωρίς τις λέξεις high level off. Θα ψηφίσουμε χωριστά. Λοιπόν, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 1 χωρίς τις λέξεις a high level of. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας χωρίς τις λέξεις αυτές. Εγκρίνεται, σαφέστατα. Είναι κανείς αντίθετος. Όχι. Τώρα, ψηφίζουμε αν θέλουμε να προσθέσουμε τις λέξεις a high level of. Θέλει κανείς να τις προσθέσουμε αυτές τις λέξεις. και είναι κατά. Εγκρίνονται και αυτοί οι όροι. Λοιπόν, περνούμε στη 12. Υπέρ, κατά εγκρίνεται. 13. Είναι συμβαστική. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 14 επίση συμβαστική. Ε, συμβατή, με συγχωρείτε. Υπέρ, κατά εγκρίνεται. Ε, εγκρίνεται και η Τροπολογία 2. 16 υπέρ κατά απορρίπτεται, 17 υπέρ κατά εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά εγκρίνεται, 20 υπέρ κατά απορρίπτεται, 23 υπέρ κατά εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά εγκρίνεται, 25 20 για παράγραφο υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 38. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30, 40 ε, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 41 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία για τη 41. 18 προς 15 εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά εγκρίνεται. 45 υπάρχει νέα παράγραφος. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 45. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 47. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 50. Δεν χρειαζόμαστε την... Δεν πρέπει να ψηφίσετε. 50-52. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58. Τελευταία ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, με συγχωρείτε, τη γνωμοδότηση στο σύνολό της. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 32. Ομόφα, λοιπόν. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε με την γνωμοδότηση του καθηγητού Κορέα Ντεκάμπος για τη σκοπιμότητα της εγωτή ομολόγων σταθερότητα. Θέλει να πει κάτι ο εισηγητής? Όχι. Προχωρούμε.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 Η Amendment 11 is compatible with είναι συμβατή με την προφορική ετροπολογία. την οποία ψηφίσαμε. Μπορούμε να την ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καλά, καλά κάναμε και ψηφίσαμε. Για να δούμε και το σύνολο. 20. Α, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 με την προφορική τροπολογία που βρίσκεται στο τέλος του καταλόγου ψηφοφοριών υπέρ κατά εγκρίνεται καταπίπτει η 14 περνούμε στην 7 του εισηγητού ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία Απορρίπτεται. Καταπίπτει και το δεύτερο μέρος. 19. Ο εισηγητής θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ, κύριε Κάμπος. Ναι, Στον κατάλογο ψηφοφοριών έχουμε ένα πλήν στην 18 και θέλουμε να γίνει συν. Τροπολογία 18. Ευχαριστώ. Για να δούμε, θα φτάσουμε στο 18 πρώτα. Λοιπόν, άντε. 19. Ε, ναι. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Αρχίζει η ηλεκτρονική, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει. Η δεκα. Όχι, την ψηφίζουμε ως προσθήκη. Υπέρ. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 16 ως προσθήκη. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 22 Υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 με χωριστή ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 10. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μια συμπληρωματική ψήφο υπέρ. 26. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψήφος για την γνωμοδότηση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία και εγκρίνεται με 23 προς 7. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κορέια Τεκάμπος. περνούμε στην εκνομοδότηση του κύριου Μπουσόη για την, ε, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θέλει να πει τίποτε ο εισηγητής. Στην πρώτη παράγραφο τροπολογία 2 De Jong. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά απορρίπτεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 υπέρ κατά Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για να είμαστε σίγουροι. Αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της χρονομοδότησης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 30 προς 1 και μία εποχή Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην έκθεση Κοφεράτη, θέλετε να πείτε κάτι κύριε Κοφεράτη. Όχι, αρχίζουμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Όχι, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Έληξε. Απορρίπτεται. Πέντε υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 ε, υπέρ ηλεκτρονικά πολύ καλή τροπολογία αυτή η εξαιρετική έληξε άλλαξε γνώμη το ΕΛΚ 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά απορρίπτεται επίση 11 υπέρ έντεκα ηλεκτρονικά. κατέληξε. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Εγκρινείται. Δεκαέξι. Πρέπει να διορθωθεί ένα μεταφραστικό λάθος εκεί. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 συμβιβαστική 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 18 πάλι θέμα μετάφρασης υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 31 κατά πίπτη εάν εγκριθούν οι συμβιβαστικέ. Συμβιβαστική 4 υπέρ Κατά. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Υπέρ 33 είπα. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι επόμενες. Τώρα η 41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 46 ηλεκτρονικά 46 έλξε απορρίπτεται 47 ηλεκτρονικά απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έληξε. συγκρίνεται 28 υπέρ μία ψήφος κατά τελική σημερινή ψηφοφορία γιατί φτάνουμε και στις 12 της κυρίας Μακκλάρκιν η γνωμοδότηση έχετε καμία δήλωση να κάνετε κυρία Μακκλάρκιν ορίστε πολύ σύντομη να ευχαριστήσω τους πάντες και πάσες που συνεργάστηκαν για να καταλήξουμε σε αυτήν την πολύ καλή γνωμοδότηση. Μάλιστα, φύγαμε. Εννέα της κυρίας Μακλάρκιν υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δέκα, διότι προηγούμενη, ναι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Του ρέπο 69 ως προσθήκη ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. 70 έχει καλυφθεί. 71 υπέρ. 71 υπέρ κατά Α, Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13 της ηγητρίας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της ηγητρίας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 της ηγητρίας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 76 ε, του κυρίου Σμιτ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά εγκρίνεται. 77 είχε εγκριθεί 11 ναι είχε εγκριθεί θα αλλάξει λοιπόν το πράγμα εδώ αυτόματα α πρέπει να την ψηφίσουμε 77 ναι, υπέρ κατά εγκρίνεται 78 υπέρ κατά εγκρίνεται 79 ηλεκτρονικά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα οι συνδυασμένες τροπολογίες. Συνδυασμένη 1 υπέρ κατά και αυτή εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά απορρίπτεται. 87 ως προσθήκη ηλεκτρονικός. Έληξε. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. 88 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ Κατά εγκρίνεται. Άρα κατά πίπτη 89. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 93 είναι προσθήκη. Ω προσθήκη λοιπόν υπέρ, υπέρ, υπέρ. 93 ως προσθήκη. Κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. πίπτη 94. 95 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε δύο καλύπτονται. 98 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 100 ως προσθήκη εκεί στην τελευταία φράση, τελευταία φράση. Υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 26 καλύπτεται. 102 καταπίπτει. 103. υπέρ. Μα εδώ ξανά υπέρ. Ε, μάλιστα. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 104. Οι 27 και 105 έχουν αυτόματα εγκριθεί. 28 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε, για να το ελέγξουμε να είμαστε σίγουροι. Έλξε. Εγκρίνεται. Με τέσσερις ψήφους διαφορά. 30. Υπέρ. 30 η ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. 9, 12 και 11 αποχές. 31 πέρ. ΠΕΡ, ΠΕΡ, Κατά εγκρίνεται πανηγυρικά. 32. Ε, κατά. Απορρίπτεται. 33. Ε, τα. Πώς, πώς, όλες μαζί. 34, 35, 36 και 37 μαζί. Υπέρ, κατά. Απορρίπτονται. 38 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά. και Α, εγκρίνεται. Τώρα στο σκεπτικό 40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 42 προφορική προσθήκη. Έτσι ε, δεν είναι, ε, δεν είναι. Λοιπόν, 42 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 3 προφορική. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 46 ως προσθήκη υπέρ, κατά εγκρίνεται. 47 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 51 του κυρίου Βαλτάσαρη υπέρ κατά εγκρίνεται 52 υπέρ Α, όχι, όχι, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά εγκρίνεται με μία ψήφο παραπάνω. 5 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. 53 γκρεκ υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 και 54 υπέρ κατά εγκρίνονται. 55 γκρεκ υπέρ κατά εγκρίνεται. 57 μπαλντάσαρε υπέρ. Περ. Τα. Εγκρίνεται. Τώρα η 56 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. 60. Μόνο εκεί που λέει για τα ποσοστά και ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 8 έχει αποσυρθεί, 65 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 66 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο, το σύνολο, ηλεκτρονικά, σύνολο. Μήπως θέλει και κανείς άλλος να ψηφίσει. Μην βγάζετε τις κάρτες σας, δεν τελειώσαμε. Εγώ σας είδα, τη βγάλατε την κάρτα σας. Εγώ δεν έληξα την ψηφοφορία ακόμα, γιατί βγάζετε τις κάρτες. Λοιπόν, τώρα λίγη. Ομοφωνία. Ευχαριστούμε την εισηγητρία. θα αφήσουμε όλο τον κόσμο σιγά σιγά να φύγει όσοι είναι να φύγουν και ο κ. Κονφεράτη είναι σύντομα εδώ για την έκθεσή του σε σχέση με τις ε, πληρωμές μέσω κινητών μέσων. Σας παρακαλώ ησυχία καθώς εγκαταλείπτε την αίθουσα. timing. Uh, um, Εξαιρετικό timing. Έχουμε προγραμματίσει πολύ καλά το χρονοδιάγραμμα. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πέντε λεπτά νωρίτερα. Η Κομισιόν είναι εδώ. Καλώς ορίζω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και το Συμβούλιο βρίσκεται εδώ. Έχουμε κάποιους παρατηρητές επίσης από την Κυπριακή Προεδρία. Έχουμε όλους τους κοιόδης εδώ. Έτσι δεν είναι. Έχουμε τον κύριο Κοφεράτη. Φυσικά ο κύριο Άρια δεν είναι εδώ. Α, όχι, είναι εδώ. Πήγατε να ξεφύγετε. Ο κύριος Σμιτ δεν είναι εδώ. Κάποιο από τους φιλελεύθερου θα μιλήσει εκ μέρου του κύριου Σμιτ. Όχι. Ο κύριος Έγκστρομ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μπίνεν είναι εδώ. Έχουμε λοιπόν απαρτία σκιωδών. Θα μιλήσουμε λοιπόν, θα συζητήσουμε για τις τροπολογίες επί της εκθεσής του κυρίου Κοφεράτη. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σιγητή ώστε να μας πει την άποψή του για τις τροπολογίες και να μας πει την άποψή του και έτσι μετά μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή την ε, γνωμοδότηση ε, για το Σεπτέμβριο. Κύριε Κοφεράτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη στους επιβιώσαντες αλλά είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε σήμερα το πρωί. Έστειλα στους σκιώδεις μετά από μια συνεδρίαση πριν από μερικές μέρες το αναθεωρημένο κείμενο των συμβιβαστικών διότι σε εκείνη τη συζήτηση όπου παρήσταν οι σκιώδεις και οι βοηθοί τους για όσους απουσίαζαν σε εκείνη τη συζήτηση λοιπόν ε, κάναμε κάποιες μικροδιορθώσεις. Νομίζω ότι κατάλαβα καλά τη συζήτηση που έλαβε χώρα, αλλά φυσικά ε, είμαι στη διάθεση όλων για τυχόν περαιτέρω παρατηρήσεις ή σχόλια που μπορεί να γίνουν επί των συμβιβασμών και αξιοποιώ την ευκαιρία, εκμετάλλευα την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, που συνεργάστηκαν εξαιρετικά και έδειξαν τεράστια υπομονή σε ένα έργο το οποίο δεν είναι πάντα απλό. Ήθελα να πω για τις ομάδες για τις οποίες δεν υπάρχει σκιώδης παρόν αλλά και για τις άλλες ότι εκτός από τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα έχουμε και άλλες μέρες σε περίπτωση λοιπόν που στα κείμενα που έχετε λάβει έχετε να κάνετε και επιπλέον παρατηρήσεις μπορείτε να μου τις στείλετε μετά από αυτή τη συζήτηση. Στις, ε, στις στο σημείο που μου φαίνεται αντικειμενικά πιο περίπλοκο και για το οποίο κατά την άποψή μου θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων. Είναι το σημείο που σχετίζεται με το συμβιβαστική G. Μια, ένα συμβιβασμό αρκετά ευρύ επειδή καλύπτει δικές μου τροπολογίες, δηλαδή τροπολογίες του κ. Σμιτ, του κ. Τριανταφυλλίδη, τη συναδέλφου Βαντούν, Μπίνεν, Σαλβίνη και του συναδέλφου Αρίας. Όπως πάντα, όταν το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ ευρύ, ενδεχομένως ε, ε, αυτή η σύνθεση που κάνουμε όλων των απόψεων να μην αντιστοιχεί ακριβώς στις συζητήσεις. Ε, ελπίζω να είμαι πιστό στα όσα μου είπαν, αλλά θα ήθελα επί αυτού του σημείου να με καθησυχάσουν και οι υπόλοιποι σκιώδεις όπως θα το επιθυμούσα. Η πτυχή που κατά την τελευταία συνεδρίαση προκάλεσε τη σημαντικότερη συζήτηση ήταν η πτυχή που σχετιζόταν με το πώς θέτουμε σταδιακά υποέλεγχο τις διατραπεζικές προμήθειες που σήμερα αποτελούν πρόβλημα διότι έχουν χαρακτήρες και διαστάσεις πολύ διαφορετικές στις εκάστοτε ευρωπαϊκές χώρες και δική μας ανησυχία είναι ότι πρέπει να επιτύχουμε όχι μόνο την εναρμόνιση αλλά και τη σταδιακή μείωση των προμηθειών χωρίς αυτό να μετακυλιστεί στους καταναλωτές, στους χρήστες δηλαδή. Γι' αυτό τον λόγο καλέσαμε την Επιτροπή να πραγματοποιήσει ήδη από το 2012 μελέτη αντικτύπου, αξιολόγηση αντικτύπου, ως σημείο αφετηρίας για την περαιτέρω, για την μετέπειτα αξιολόγηση. Όσον αφορά τις υπόλοιπου συμβιβασμού αλλά και τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν, πιστεύω ότι υπάρχει διάθεση να προχωρήσουμε προς ε, την κατεύθυνση που επιθυμώ ώστε να επεκτείνουμε αυτούς τους όρους πληρωμής ε, με τρόπο ωστόσο όσο το δυνατόν καλύτερο, δηλαδή έναν τρόπο που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εγγύηση για τους χρήστες, τους καταναλωτές να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε διαδικασίες χωρίς επιζήμια αποτελέσματα από αυτή την υιοθέτηση. Ουσιαστικά οι πολίτες είναι ιδιαίτερα διατεθειμένοι να δεχθούν τέτοιες ε, ε, διατάξεις, αλλά το πρόβλημα μπορεί να είναι αυτή η έλλειψη γνώσης αυτής της διαδικασίας, η έλλειψη φυσικής επαφής μεταξύ καταναλωτή και τράπεζας ή οποιοδήποτε διάμεσου κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες δυσκολίες ή και σε ζημίες για τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, έχουμε τα άτομα μεγαλύτερη ηλικία που είναι ελάχιστα εξοικειωμένα με ε, την ορολογία αυτή και αυτές τις τεχνολογίες και ε, ε, είναι πιο επιφυλακτικοί στη χρήση αυτών των μέσων. Θεωρώ ότι εδώ δίνουμε μια ικανοποιητική απάντηση κυρίως ε, χαρίς τη συμβουλή της τροπολογίας και την εργασία των σκιωδών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για επέκταση αυτών των διαδικασιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς ε, όφελος των καταναλωτών που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πιο γρήγορο, πιο ε, διαχειρίσιμο, πιο εύκολα διαχειρίσιμο μέσο. Επίσης αυτές οι διαδικασίες θα επιτρέψουν την απαλυφή μελανών σημείων, ασαφών σημείων που αντικειμενικά κλασικά προσελκύουν ε, οποιονδήποτε κινείται παράνομα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια δυνατότητα καλύτερης υπηρεσίας προς τους χρήστες, μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο για τους χρήστες όσο και για ε, τους ε, δικαιούχους των πληρωμών τους παραλήπτες των πληρωμών και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια διαδικασία αυτοματισμού που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που εξάλλου είναι και στόχοι αυτής της Επιτροπής. Αυτό θα παίξει το ρόλο. Σας ζητώ λοιπόν να μου δώσετε προς τα σχόλια και εάν δεν μπορείτε να τα δώσετε εδώ στείλτε μου τα πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες για αυτό το έγγραφο και μάλλον αφού ολοκληρωθούν οι εργασίε αυτή τη επιτροπή, στείλτε μου οποιασδήποτε σκέψει και σκέψει για την συμβιβαστική G που ήταν η πιο ευρεία φύση ε, συμβιβαστική. Και ξανά ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ που αναφέρατε αυτά τα σημεία. Δίνω το λόγο τώρα στους σκιώδεις ξεκινώντας από τον κύριο Άριας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη, τον Σέρχιο, διότι ανα πάσα στιγμή ήταν στη διάθεση των σχεδόν εισηγητών εμού αυτοπροσώπους. Και θα πρέπει να πω ότι τώρα που μιλούμε για το σχέδιο γνωμοδότησης και για τα θέματα τα οποία είχαμε σε σχέση με ε, αντιφατικά θέματα που θα μπορούσαν να προκύψουν, πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνήσαμε σε όλα τα θέματα που τέθηκαν και για το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών μας. Η θέση της ομάδας μου λοιπόν είναι η εξής, ότι καταρχήν, όπως και ο κύριος Κοφεράτη γνωρίζει πολύ καλά, Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα των διαφόρων ε, διαπραγματεύσεων και με τα αποτελέσματα γενικότερα, άρα σχεδόν συμφωνούμε με όλο το περιεχόμενο της γνωμοδότησης έτσι όπως έχει διατυπωθεί. Αυτό ήθελα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Σμίτ, ο κύριος, κύριος Σμίτ, κύριος Μπίλαν, ποιος θέλει πρώτος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή. που συμπεριέλαβε όλες τις τροπολογίες σχετικές. Εγώ κατέθεσα μία τροπολογία, την 25, με τον συνάδελφο Ανταμτούν και πρέπει να πω ότι χαίρομαι με τις συμβιβαστικές τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν τις περισσότερες από αυτές θα θέλαμε να έχουν συμπεριληφθεί και βεβαίως με ικανοποιεί και η ε, αξιολόγηση επιπτώσεων που θα παρουσιαστεί και τα, αυτά τα οποία προβλέπονται. Κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ. το πρωί έτρεχα σε διάφορες επιτροπές, γι' αυτό καθυστέρησα. Νομίζω όμως ότι καταλήξαμε σε πολύ σωστό συμβιβασμό και ευχαριστώ όλους που έκαναν την προσπάθεια και τον εισηγητή ιδιαίτερα. Το έχω ξαναπεί ότι το θέμα είναι σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ περισσότερη ευρωπαϊκή εναρμόνιση για αυτή την αγορά. Επίσης σας ευχαριστώ γιατί συμπεριλάβατε τις συστάσεις μου ιδιαίτερα εκείνη που κάνει λόγο για σημεία επαφής. Γενικά λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και ελπίζω το Σεπτέμβριο να εγκριθεί άνετα και να υπάρξει ευρία ψηφία. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά τον εισηγητή και ελπίζω η καλή αυτή συνεργασία να συνεχιστεί και στο μέλλον. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κανένα άλλο μέλος που να μην είναι σκιώδης. Ο κύριος Χάιλαντ μήπως θέλει να πει κάτι για τις τροπολογίες και μετά ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτώντας όλες τις τροπολογίες που μελέτησα, αυτό που εκτιμάμε ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει αυτή η έκκληση για περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς μέσω των γεννητών πληρωμών και γίνεται έκκληση για ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Γνωρίζουμε ότι η ενοποίηση των πληρωμών είναι εξαιρετικά σημαντική για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για την ψηφιακή ενιαία αγορά και αυτό αποτυπώνεται ξανά και στις ε, τροπολογίες ε, Είμαστε λοιπόν υπέρ των περισσότερων τροπολογιών που είδαμε. Για να επανέλθουμε στο σημείο κλειδί, τις προμήθειες αυτές, τις διατραπεκές προμήθειες, αυτό που μάθαμε από την δημόσια διαβούλευση ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα μεταξύ ενδιαφορομένων. Υπάρχει αυτή η διχογνωμία μεταξύ της πλευράς προσφοράς και ζήτησης της αγοράς και εξετάζουμε και τις δύο απόψει ε, σε αυτό το στάδιο αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορά των προμηθειών αυτών μπορεί να αποτελέσει φραγμό για την ενιαία αγορά και εξετάζουμε αυτά τα τέλη για να δούμε σε ποιο βαθμό αποτελούν φραγμό στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τις πληρωμές με κάρτες αλλά και για τις ε, υπηρεσίες που παρέχουν οι παροχές καρτών σε λιανοπολιτές. Εξετάζοντας όλα αυτά θα προβούμε σε ανάλυση αντικτύπου. Να σας υπενθυμίσω διότι πολλές τροπολογίες που δεν συζήτησαμε σήμερα το πρωί αφορούν και την προστασία των καταναλωτών. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή τη στιγμή αναθεωρούμε την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και αναφέρεται ότι κάποια από τα μέτρα follow-up ε, που υπάρχουν στο πράσινο βίβλο μπορούν να ε, εξεταστούν μέσω αυτής της αναθεώρησης τώρα της οδηγίας αυτής και θα κάνουμε μια ανακοίνωση πριν το τέλος του καλοκαιριού για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ποια είναι οι τομείς προτεραιότητα στην Πράσινη Βίβλο και πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much. I think, um, Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ανυπομονούμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εξέταση. Θέλατε να πείτε κάτι κύριε Κομφεράτη, να ολοκληρώσετε. Ναι, γρήγορα θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τους συναδέλφους μου για τη δουλειά τους και για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή τη συζήτηση διότι και η στάση και το πνεύμα πιστεύω μετρούν πολύ όταν έχουμε να κάνουμε με σημαντικά και ταυτόχρονα ευαίσθητα και πολύπλοκα θέματα. Μια σύσταση έχω να κάνω στην Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις δυσκολίες. Εξάλλου, τις ίδιες δυσκολίες ε, αντιλαμβανόμαστε και εμείς όσον αφορά τις δύο αυτές διαφορετικές τάσεις για τις διατραπεζικές ε, προμήθειες ε, τους χρήστες αφενός και της τράπεζες αφετέρου. Μην υποτιμάτε ωστόσο την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει η Επιτροπή ΙΜΚΟ και όλες τις συνιστώσεις για να καταφέρουμε να διατυπώσουμε το κείμενο με τρόπο ισορροπημένο. Δεν ήταν κάτι το εύκολο. Ιδιαίτερα διότι ορισμένε φορέ όσοι κάνουν αυτήν εδώ τη δουλειά μπορεί να κληθούν να λάβουν θέση υπέρ του ενός υπέρ του άλλου. Πιστεύω ότι η διατύπωση στην οποία έχουμε καταλήξει είναι ικανοποιητική, δείχνει, Καταδείχνει μια διαδρομή που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά δίνει μια διαδρομή αρκετά θετική πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Okay, well, thank you very much. Uh, anyway, we have until... Πολύ καλά, σας ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε στις 6 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε υπάρχει χρόνος για περαιτέρω συμβιβαστικές τροπολογίες μεταξύ εισηγητού και σκιωδών και αργότερα χρονικά θα ψηφίσει η οίκον που είναι υπεύθυνη της ουσίας την εκθεσή της. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε για σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 3 σήμερα το απόγευμα για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας θα καλωσορίσουμε τον ε, Προεδρεύοντα, τον ε, Κύπριο Υπουργό Υπεύθυνο για Εμπόριο, Βιομηχανία και Τουρισμό. Τώρα θα έχουμε γεύμα μαζί του, Πρόεδρος και συντονιστές. Μετά θα ψηφίσουμε τις ε, την, θα, θα συζητήσουμε έκθεση De Jong, μετά ψηφοφορία των εκθέσεων Ρόιτοβα και οι συντονιστές και κλεινό των θυρών θα συνεδριάσουν από τις 5 και 4. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλή σας όρεξη.